Ladies and gentlemen, good morning once again. Σας καλημερίζω και πάλι. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι. Ας επαναλάβουμε τις εργασίες μας, τις εργασίες της Επιτροπής. First Το πρώτο θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω και να σας πω ότι σήμερα το πρωί χρειαζόσαστε την κάρτα σας για να ψηφίσετε. Και επίσης θα ήθελα να σας μιλήσω για τις αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν λίγη ώρα πριν. Η κυρία Φεράρα διορίστηκε η για το νέο αίτημα άρσης της ασυλίας του κυρίου Σπάσκιχ. Ο κύριος Χρυσόγονος διορίστηκε εισηγητής για την ε, άρση της ασυλίας του κυρίου Μαρίνιου Πίντου συμφωνήθηκε να γίνει μια κοινή ακρόαση Γιούρι και Ίντα για το TTIP, για τις ρυθμιστικές ε, πτυχές και την ε, διατησία διαφορών μέσα στα πλαίσια του TTIP το 2015. To hold a hearing only of our jury committee στις 19, 19 μέχρι 22 Ιανουαρίου και να ασχοληθούμε την ίδια μέρα ε, με την επίλυση διαφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΙΠΑ. Επίσης, η αντιπροσωπεία στη Λετωνία θα γίνει μόνο με λετωνικά και αγγλικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις λοιπόν των συντονιστών. Και συνεχίζουμε με το σημείο 14, τροποποίηση του κανονισμού του συμβουλιου 1346 1446-2000 περί διαδικασιών αφαιρεγγιότητας. Ο κύριος Βιέφκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά πριν από την ψηφοφορία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία επί του κανονισμού αυτού. Οι διαδικασίες αφαιρεγγιότητας είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Μιλάμε για επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφανθεί επί του θέματος για να υπάρχει σωστή μεταχείριση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο δεν ήταν απλές, αλλά είχαμε σωστή προσέγγιση στον τριμερή διάλογο και έτσι φτάσαμε σε συνένεση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι ως Κοινοβούλιο γιατί προωθήσαμε τις θέσεις μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και τους συνεργάτες από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ωραία. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Βλέπουμε ότι είμαστε υπεράριθμοι στην ψηφοφορία. Θα μπορούσαν οι πολιτικές ομάδες να ελέγξουν παρακαλώ. Κατά πόσο αυτοί που ψηφίζουν είναι ή δεν είναι υπεράριθμοι. Δείτε το θέμα σε κάθε πολιτική ομάδα. Ψηφίζουμε και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Σύμφωνα με τη γραμματεία, 21 μπορούν να ψηφίσουν και έχουμε 23 που ψηφίζουν. Άρα υπάρχει κάποιο θέμα. Εντάξει τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια έχουμε το 15 αναφορές σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόορης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία. Ε, ψηφίζουμε διανατάσεως της χειρός. Υπέρ παρακαλώ. κατά αποχές ουδεμία εγκρίνεται ευχαριστώ πολύ Δεκαέξι, το 16 έχει αναβληθεί. 17 on block μέχρι το 23. με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε 23 ε, ψηφίσαντες. Η σοσιαλιστική ομάδα θα πρέπει να έχει 6 που να ψηφίσουν, τώρα έχει 8. Έχει δύο υπεράριθμους. εντάξει με τους πράσινους. Παρ' όλα αυτά έχουμε 23 ε, ψηφίσαντες. Το ΕΛΚ έλεγξε. Σας παρακαλώ ποιος ή όποια δεν πρέπει να ψηφίσει μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα σας από το μηχάνημα. Τώρα είμαστε εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνονται οι εκθέσεις αυτές. 24. Το λόγο έχει η συγγήτρια κυρία Ρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση για την ε, εναρμόνιση της οδηγίας InfoSoc και ορισμένα δικαιώματα ε, διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να σας δώσω ορισμένες προθεσμίες και να σας πω πώς εξελίχθηκε η έκθεση. Περιμένω ένα λεπτό. So, uh, the InfoSoc Directive... Η οδηγία InfoSoc εγκρίθηκε 13 χρόνια πριν για να εναρμονιστούν ορισμένα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και για να ανταποκριθούμε στις αλλαγές στην ψηφιακή κοινωνία και περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η οδηγία InfoSoc έχει επιτύχει το στόχο της εναρμόνισης έμπρακτα στα διάφορα κράτη-μέλη και ποια νομικά βήματα θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα σε σχέση με το θέμα της εδαφικότητας των πνευματικών δικαιωμάτων. Πέρα από το θέμα του κατά πόσο αυτό το μέσο εναρμόνει σε ορισμένες πτυχές των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει σε σχέση με την αρχική διατύπωση της οδηγίας InfoSoc του 2001. Ορισμένες λύσεις είναι αναχρονιστικές σε σχέση με τους κανόνες που διέπουν τις ε, βιβλιοθήκες και την πρόσβαση αρχιακού υλικού ή υλικού βιβλιοθήκης σε περίπτωση ανάγνωσης σε βιβλιοθήκες. Η οδηγία μιλά για τεχνολογίες τύπου CD-ROM που είναι αναχρονιστικές και τα τελευταία 13 χρόνια έχουν ανακύψει νέες χρήσεις που ίσως δημιουργούν προβλήματα ως προς την εφαρμογή της οδηγίας InfoSoc. Ποιες ε, ομάδες ε, πλήττονται από την ε, εφαρμογή της οδηγίας λοιπόν InfoSoc και ποια προβλήματα υπάρχουν και μας ανέφεραν στις διαβουλεύσεις, ιδιαίτερα στα προσκόμματα, ως προς τα προσκόμματα για καινοτόμα στοιχεία που έχουν μπει στην αγορά ή να είμαστε σε θέση να δώσουμε τις σωστές αμοιβέ σε αυτούς που προβάλλουν αυτά τα καινοτόμα στοιχεία ή στους χρήστες. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά μας, θα σας υποβάλω ένα πρώτο σχέδιο κατά τα μέσα του Ιανουαρίου και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η Επιτροπή για την ε, υποβολή μιας πρότασης νομοθετικού περιεχομένου για τη μεταρρύθμιση ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάτι που θα ανακύψει το καλοκαίρι του 2015 και ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει νέα στοιχεία για αυτή την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως θα ανακύψουν το 2015. Για τις τροπολογίες θα υποβληθούν το Φεβρουάριο και ίσως και την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα έτσι ώστε να ψηφίσουμε στις 24 Μαρτίου στη Γιούρη και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Το EPRS ασχολείται με, την, με τον ευρύτερο αντίκτυπο ως προς το κόρπους των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο και θα δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος όλων των οδηγιών που ασχολούνται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Και στη συνέχεια θα έχουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου από την Επιτροπή το επόμενο έτος. Η Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το EPRS, θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και θα δούμε ποιες είναι οι διάφορες προκλήσεις της οδηγίας InfoSoc στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα. Η κυρία Χάνιμπο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την κυρία Ρέντα για αυτή την αναλυτική παρουσίαση. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση, αυτή η επανεξέταση της εφαρμογής της νομοθεσίας γιατί αλλάζει ταχύτατα η κατάσταση στον τομέα αυτό και είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όταν νομοθετούμε γιατί μόνο λίγα χρόνια έχουν περάσει από το 2001 και έχουν γίνει τρομερές αλλαγές. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά βιβλία όπως το Kindle δεν υπήρχαν τότε. Και στην, στον τομέα της μουσικής έχουν γίνει τρομερές αλλαγές. Όλοι ακούνε τώρα μουσική μέσω του ίντερνετ και κατεβάζουν ε, κομμάτια μουσικής, δεν αγοράζουν CD εντελώς διαφορετική κατάσταση. Είναι λοιπόν ε, όντως πολύ απαιτητική η κατάσταση και πολύ δυσχερής η προσπάθεια να νομοθετήσουμε. Αυτή λοιπόν ε, η επισκόπηση του πώς εφαρμόστηκε η προηγούμενη νομοθεσία θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε καλύτερα ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αλλά υπάρχουν μερικές σημαντικές αρχές τις οποίες πρέπει να έχουμε υπόψη όσο θα εξετάζουμε την εφαρμογή της προηγούμενης οδηγίας και για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και ένα θέμα πολύ βασικό, μοιάζει προφανές, αλλά πρέπει να υποθεί, πρέπει να υπάρχει σωστή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η προστασία δεν θα γράφονται βιβλία, δεν θα γράφεται μουσική δεν θα έχουμε τα τηλεοπτικά προγράμματα που θέλουμε. Εάν δεν προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα για να βοηθήσουμε τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, όλους τους άλλους, όλους που είναι στα παρασκήνια και βοηθάνε να καταλήξουμε σε ένα καλλιτεχνικό προϊόν, σε ένα βιβλίο, δεν θα πληρωθούν όλοι αυτοί. Άρα θα φύγουν από τον τομέα αυτό. Μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό, αλλά έτσι γίνεται. Αυτό συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό κάτι πολύ σωστό που ανέφερε η κυρία Ρέντα, που πρέπει να λάβουμε υπόψη ιδίως για το μέλλον, είναι η εδαφικότητα. Γιατί νομίζω ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Και υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις στον κλάδο για το θέμα αυτό. Όσοι εργάζονται στα οπτικοακουστικά έχουν πολύ διαφορετική άποψη για αυτό το θέμα εδαφικότητας από τους μουσικούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίω πρέπει να παρακολουθούμε την τεχνολογική πρόοδο, αλλά αυτή πρέπει να είναι η βασική μας αρχή. Πρέπει να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κομοντίνη. Ως κοιόδης ε, του ΕΛΚΑ προσβλέπω στη συνεργασία για το θέμα αυτό Συμφωνώ στα περισσότερα που αναφέρατε ότι η έκθεση πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της διαρκώς μεταβαλλόμενης τεχνολογίας μέσω των οποίων ε, έχουν πρόσβαση οι χρήστες ε, στα προϊόντα αυτών. Και το ερώτημα που τίθεται είναι μπορούμε να εγκρίνουμε ένα νομοθέτημα που να μπορέσει να έχει έννοια εφαρμογή του σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο τοπίο. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε κάποιες αρχές. Καταλαβαίνουμε ότι η έρευνα και η καινοτομία θα συνεχίσουν να ε, βοηθούν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οποιοδήποτε νομοθέτημα πρέπει να βοηθήσει λοιπόν την ιδιωτική επένδυση στην έρευνα και καινοτομία, να προστατεύει τους δημιουργούς, αλλά παράλληλα πρέπει να φροντίζει οι υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες για τους χρήστες. Οποιαδήποτε πρόταση θα υποβάλουμε μέσω της έκθεσης αυτής πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συμβαδίζει με την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία της πληροφορίας. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, νοοτροπία των χρηστών. Γιατί και οι δικές τους ε, απόψεις για το πώς πρέπει να υπάρχει πρόσβαση μέσω του ίντερνετ ε, στα προϊόντα αυτά αλλάζουν. Και πιστεύω ότι κάτι άλλο που πρέπει να είναι στη βάση της έκθεσης είναι πώς θα επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των κινήτρων για τους δημιουργούς, δηλαδή να προστατεύουμε αυτούς ε, που έχουν τις πρωτότυπες ιδέες και να προστατεύουμε και τις εταιρείες που μας χορηγούν αυτά τα προϊόντα και να σεβόμεθα επίσης και τις συνήθειες και τη στάση των ε, χρηστών, των καταναλωτών. Εδώ θα είναι η ουσία, αυτή η ισορροπία θα είναι η ουσία των προτάσεων που θα πρέπει να υποβάλουμε. Προσβλέπω όμως σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Καβαντά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι και η κυρία Χάνιμπαλ συγκεκριμένα. Δεν θα πρέπει να διαπράξουμε ένα ιστορικό και καταστροφικό σφάλμα ή να θεωρήσουμε ότι ο εξυγχρονισμός των ζητημάτων πρόσβασης σε, ε, σε πολιτιστικά έργα ε, θα δημιουργήσει η οικονομία του πολιτισμού. Θέλω να επιμείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, στο ότι είμαστε σε ένα μετέχμιο. Χωρίς οικονομία του πολιτισμού δεν υπάρχει πολιτισμός. Μπορεί κάποιος ε, ε, στο δικό του χώρο κάτι να φτιάξει και να δούμε ένα θέαμα σε μια πλατεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα όμως είναι ότι θα ανοίγαμε διάπλατα τις πόρτες ε, σε μια δεσπόζουσα βιομηχανία, την αγγλοσαξονική και για να μην πω συγκεκριμένα την αμερικανική βιομηχανία, γιατί θεωρώ ότι οι Βρετανοί εντάσσονται στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος, μια και καλυμμένη ε, προέλαση αν θέλετε, γιατί μας μιλάνε για πρόσβαση στην αγορά. Υπάρχει ε, πρόσβαση στην αγορά των προκυπευτικών. Μπορεί κανείς να πάρει πατάτες ε, ή κάποιο άλλο προκυπευτικό χωρίς να πληρώσει. Όχι. Ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν κάποιες ιδέες ε, που εμείς όμως δεν τις βρίσκουμε ίσως, δεν είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Αυτό που θέλουμε είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτισμών, αν θέλετε, αναχώρα, γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της πολιτισμό, αλλά σε ένα υπηρετικό σύνολο, όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένο και βέβαια με εύκολη πρόσβαση. Όμως, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος εδώ και το τονίζω, γιατί δεν θέλω να το υποβαθμίσουμε και το βλέπουμε πολύ ε, καιρό ότι κάπως και καλυμμένα πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση λέγοντας ότι όλα πρέπει να είναι ελεύθερα και δωρεάν όμως όχι. Στο δεύτερο θα πω όχι γιατί αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν όλε αυτές τις υπηρεσίε του διαδικτύου δεν το παίρνουν από το σούπερ μάρκετ τσάμπα, πηγαίνουν και πληρώνουν και τον αγοράζουν τον υπολογιστή. Είναι ένα άκρο πολιτικό ζήτημα τόσο πολύ που αφορά το ίδιο το δημοκρατικό σύστημα στην πράξη. Έχουμε τα πολιτικά συστήματα των πολιτισμών, αλλά όχι το αντίστροφο. Δεν έχουμε πολιτικό πολιτισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων. Έχουμε τα πολιτικά συστήματα, ε, την αρμονική συμβίωση, έχουμε κάποιους νόμους που βασίζονται ε, στο πολιτισμικό μας υπόβαθρο. Και πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί γιατί μας παρακολουθούν. Στην Ευρώπη, και θα ολοκληρώσω με αυτό, έχουμε δύο δυνατότητες. Είτε ευθυγράμμιση περιεχομένου στο δίκτυο Και το δεύτερο είναι να θεωρήσουμε ότι Είμαστε σαν αυτοί που είχαν πετρέλαιο στο υπέδαφος μεταξύ των δύο ε, παγκόσμιων πολέμων. Αλλά αυτοί που είχαν τους αγωγούς ήταν αυτοί που θα πλούτιζαν τελικά των δικτύων. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μια φορολογική εναρμόνιση για να προωθηθεί η αξία του πολιτισμού. Ευχαριστώ. Merci ε, Σας ευχαριστώ, κύριος Κέστερ. Είναι προφανές ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί το copyright. Είναι βασική προϋπόθεση για να προωθήσουμε τη δημιουργία πολιτιστικών αγαθών. Θέλω να αναφερθώ στα εξή σημεία για την επερχόμενη συζήτηση. Πιστεύω ότι στον τομέα του πολιτισμού έχουμε τέσσερις κύριους παρεμβαίνοντες, τους δημιουργούς, τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους χρήστες ή καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή οι έμποροι έχουν ε, την κυρίαρχη θέση και αυτοί εποφελούνται από την ψηφιοποίηση της ε, ε, διάδοσης των πολιτιστικών προϊόντων. Πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη περισσότερο τους δημιουργούς. Όπως είπε και η κυρία Χάνιμπουλ, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν τα πολιτιστικά έργα και πρέπει να τους βοηθήσουμε μέσω εξυγχρονισμού του κανονισμού των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστά εξορροπημένη σχέση μεταξύ των δημιουργών, των παραγωγών, των ε, παρόχων των υπηρεσιών και των χρηστών. Αυτό είναι το κύριο καθήκον μας. Θέλουμε λοιπόν έναν πολιτιστικό κλάδο και για αυτό το λόγο πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να αποφύγουμε τις ε, ε, απομιμήσεις και την πειρατεία. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό, να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα της πειρατείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια των συναδέλφων. Θα ήθελα όμως να τονίσω μια πτυχή. Στις μέρες μας ο πολιτισμός δεν είναι μια ε, περιορισμένη αποκλειστική δραστηριότητα που θα πρέπει να την προστατεύσουμε για πολλούς λόγους. Ή παραδείγματος για να διατηρήσουμε την εθνική ταυτότητα, γιατί ο πολιτισμός έχει γίνει πλήρη οικονομίας. Παράγονται θέσεις εργασίας. Απασχόληση. Έχουμε λοιπόν ε, την ε, πολιτιστική βιομηχανία. Και αν υπάρξει ε, ναρμόνιση μεν στην αγορά, αλλά απ' την άλλη έχουμε κατακαιρματισμό σε 28 υποτομείς στο διαδίκτυο, μπορεί να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να επεκτείνουμε την εδαφικότητα στην Ευρωπαϊκή Νοσιακή Επικράτεια. Θα πρέπει δηλαδή να εναρμονιστούν ε, τα εδαφικά δικαιώματα. Ιδάλλως η ψηφιακή αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μιλάω για βιβλία μόνο, για ηχογραφήσεις, μουσική, αλλά και για τις ταμπλέτες, ε, τα φωτοαντιγραφικά ή άλλα μηχανήματα, τα Xerox, όπου μπορούμε, μπορεί κανείς να μεταφορτώσει κάτι, να κατεβάσει ε, ή να αντιγράψει, γιατί η ταμπλέτα μου μπορεί να αντιγραψει γιατι η ταμπλετα μπορει να χρησιμοποιηθει για αντιγράφη περιεχομένου, άρα εντάσσεται στο δίκαιο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, άρα υπάρχει σχέση με τις οικονομικές εξέλιξεις και την αγορά. Άρα είναι ευρύτερο το θέμα, δεν αφορά μόνο τη νοματική ιδιοκτησία, που δεν συμβατεί με τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε νόμους για τα του δημιουργού, που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Δεν λειτουργεί όμως αυτό το σύστημα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η παράνομη αλλά ιδιαίτερα αυθυρή ε, κουλτούρα της αντιγραφής. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα του δημιουργού και είναι σημαντικό αυτό το καθήκον. Και σε ό,τι αφορά και τι ενημερωτικέ εκστρατείε. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Κύριο Μαρίνιο Πίντου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το ζήτημα αυτό έχω τις δικές μου σκέψεις. σύμφωνο με τις προϋποθέσεις μιας οικονομίας του πολιτισμού, αλλά έχω ορισμένε επιφυλάξεις. Γιατί επικρατεί μια στάση, ας το πω, των ζηλωτών γύρω από αυτό το θέμα δηλαδή στάση άκρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως προς την πνευματική εργασία ο Δάντης, ο Πετράρχης, ο Καμόης, ο Ρούμπενς, ο Μπαχ, ο ε, Μπετόβεν και ο Φιδίας στην ε, αρχαία Ελλάδα δεν είχαν ε, κάποια αμοιβή για τα πνευματικά τους δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχει ένας μερκαντιλισμός του πολιτισμού που δεν είναι σωστός. Άρα οι μεγάλες μάζες των καταναλωτών βρίσκονται πολύ μακριά, θα απομακρυνθούν από αυτά τα πνευματικά έργα. Γιατί αν λαμβάνουμε καθερά οικονομικά μέτρα και δημιουργούμε προσκόμματα στα ευεργετικά δικαιώματα χρήσης, τότε κανείς δεν θα ασχολείται με την καλή μουσική και τα καλά βιβλία, δηλαδή θα παραμείνουν στις ελίτ. Το διαδίκτυο άνοιξε διάπλατα τις πόρτες και τους ορίζοντες έτσι ώστε αυτά τα έργα να είναι έργα των μαζών. Δηλαδή ο μέσος άνθρωπος να είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος και να μπορεί να διαβάσει, να ακούει καλή μουσική και ούτω καθεξής. Μέσω της ψηφιακής ανάγνωσης μπορεί να διαβάζει εκπληκτικά έργα, τα οποία δεν μπορούσε να διαβάζει σε μια εποχή που έπρεπε να έχεις χρήματα για να μπορέσεις να διαβάσεις αυτά τα μεγάλα έργα. Άρα, δεν συμφωνώ με τον κύριο Καβαντά όταν συγκρίνει ένα πολιτιστικό έργο με τα οποροκυπευτικά. Το πνευματικό έργο μπαίνει στο σπίτι μας διαφορετικά και δεν θα πρέπει να απολοποιούμε τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό που αλλάζει τον κόσμο, τον πλανήτη και την ανθρωπότητα, καθώς και τον ίδιο τον πολιτισμό. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε το καινούριο. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στα καλλιτεχνικά και πνευματικά έργα στο διαδίκτυο και να μην είναι προνόμιο των ελίτ. Αυτή η κοινωνικοποίηση του πολιτισμού είναι ένα θετικό έργο το οποίο δεν μπορούμε να καταστρέψουμε με μία μερκαντιλιστική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών. Τώρα η πειρατεία είναι κάτι το διαφορετικό που χρησιμοποιούν δηλαδή αυτά τα έργα για προσωπικό τους πλουτισμό. Αλλά θέλω να ακούω ό, τους πάντες σπίτι μου, από τον Μόρισον μέχρι τον Μπετόβεν μέχρι τον Βάγνερ. Γιατί αγοράζω έναν υπολογιστή και έναν εξοπλισμό για να έχω αυτή την πρόσβαση. Πρόκειται για ένα ανυπολόγιστο αγαθό στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ολόκληρος ο κόσμος σε αυτά τα εξαιρετικά καλλιτεχνικά έργα μπορούμε να δούμε ωραίους πίνακες ή να διαβάσουμε καλλιτεχνικά έργα στα οποία δεν θα είχαμε πρόσβαση διαφορετικά. Ε, thank you, Mrs. Merci, euh, ευχαριστώ πολύ. Πανέρχομαι στο κατά πόσο τα πολιτιστικά αγαθά έχουν οικονομική αξία ή όχι. Αν δούμε τα ποσά ε, που προκύπτουν από τις ε, συναλλαγές με πολιτιστικά αγαθά διαπιστώνουμε ότι έχουν οικονομική αξία τα πολιτιστικά αγαθά. Βέβαια δεν θα πρέπει αυτό το λόγο να τα θεωρήσουμε ως ένα οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα. Αιτιολογεί όμως αυτό το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν καμία οικονομική αξία και μπορούμε να τα έχουμε στη διάθεσή μας εντελώς δωρεάν. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε λοιπόν ε, και όταν εξετάζουμε αυτό το ζήτημα και στο ε, καθεστώς που αποδίδουμε στα πολιτιστικά αγαθά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την πολιτιστική διανοητική αξία αυτών των αγαθών. Υπάρχουν πολιτιστικά αγαθά που σίγουρα πλέον ε, είναι κοινή κληρονομιά, άρα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. Η δημιουργία όμως δεν είναι μόνο τα έργα του παρελθόντος, αλλά είναι μια διαδικασία που είναι σε συνεχή εξέλιξη. Και στην Ευρώπη έχουμε σήμερα την τύχη να έχουμε πολύ ανθίζουσα πολιτιστική παραγωγή και βιομηχανία. Υπάρχουν και κάποιοι μεσάζονται σήμερα, οι οποίοι ε, βγάζουν, έχουν πολύ μεγάλο τζίρο, ε, από τα πολιτιστικά αγαθά, δεν θα πρέπει όμως να διαρρήξουμε τον πολιτιστικό ιστό αυτόν τον τόσο πλούσιο, αντίθετα να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή του. Αυτός είναι ο στόχος. Thank you very much. Uh, this... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν έχω άλλους στο κατάλογο μιλτών, οπότε να δώσω και πάλι το λόγο <clears throat> στην κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ τους αδέλφους για τις πολλές σημαντικές παρατηρήσεις τους. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε η σκιώδη συγκήτρια κυρία Χάνιμπο ότι πρέπει να υπάρχουν τα σωστά κίνητρα για τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς να συνεχίσουν να δημιουργούν και χαίρομαι πολύ που η Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για να δούμε πώς μπορούν να αποδώσουν τα κίνητρα. Κάναμε και αυτή την ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας με ειδικού που ήδη μας έδωσε μερικές ιδέες. Στην ίδια κατεύθυνση συμφωνώ με τους συναδέλφους Καβαντά και άλλους που είπαν ότι παράλληλα πρέπει να διασφαλίσουμε πρόσβαση των χρηστών στα πολιτιστικά αγαθά αλλά και αμοιβή για τους ε, δημιουργούς. Ο κύριος Κώστα στην ίδια κατεύθυνση είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μεσάζοντες είναι σε θέση ισχύω έναντι των δημιουργών. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική θέση των ε, δημιουργών έναντι των ε, διαμέσων δηλαδή οι εταιρείε συλλογή ε, πνευματικών δικαιωμάτων να διανέμουν για παράδειγμα τα ποσά που συλλέγουν πραγματικά στους δημιουργούς. Και βεβαίως πρέπει να είναι εύκολη και η καταχώρηση των έργων. Όποιος θέλει δηλαδή να χρησιμοποιήσει ένα έργο να μπορεί εύκολα να δει πού είναι τα πνευματικά δικαιώματα, ποιος τα κατέχει για να, τα, για να μπορέσει να πληρώσει. Βεβαίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, έχει μιλήσει για την ανοιχτή πρόσβαση στα πλαίσια του Horizon 2020, αλλά βεβαίως έχουμε ακόμη θέματα σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα για να υπάρχει δυνατότητα χρήσης ε, των κειμένων για συλλογή στοιχείων και για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, την ανταγωνιστικότητα των επιχείρησεών μας που πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν στοιχεία με εύκολο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και να επανεξετάσουμε και την οδηγία για τις βάσεις δεδομένων. Αλλά δεν είναι θέμα απλώς προσαρμογής ε, των πνευματικών δικαιωμάτων στις τεχνολογικές αλλαγές, Πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει την ψηφιακή αγορά. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε τώρα για την εδαφικότητα είναι ότι έρχεται σε αντίθεση με τη διαφάνεια του νομικού συστήματος. Για να έχουμε λοιπόν καλύτερα νομοθετήματα πρέπει να είναι σαφές για τους χρήστες του ίντερνετ ε, τι δικαιούνται να κάνουν και τι δεν είναι νόμιμο. Ευχαριστώ λοιπόν ε, για τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις σας και προσβλέπω στη συνεργασία ε, μεταξύ όλων ημών για αυτή την έκθεση. Ο κύριος Καβαντά θέλει κάτι να πει ακόμη. Ναι, με συγχωρείτε. Να σας ενημερώσω για το εξής η ομάδα εργασίας για τα, για τα πνευματικά δικαιώματα θα αρχίσει εργασίες του 17 ε, Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο παρουσία του Επιτρόπου Έτιγκα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να περάσουμε στο 25. Και να δώσω το λόγο στην κυρία Αγωζιέ. Ευχαριστώ. θα σας υποβάλω την ε, πρόταση έκθεσης ε, πρωτοβουλίας σε απάντηση στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την επέκταση των γεωγραφικών ενδείξεων σε μη γεωργικά προϊόντα. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά προϊόντα που σχετίζονται με διαφορετικές ε, μέθοδους παραγωγής προϊόντα από τη Σκοτία, μάρμαρο της Καράρας και ούτω καθεξής που έχουν σχέση με τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης και επειδή είναι απότοκα αυτής της ε, ε, τεχνογνωσίας και ποιοτικά προϊόντα και επειδή εκπροσωπούν ένα συγκεκριμένο πολιτισμό είναι θύματα αυτής της ε, γνώσεις που έχουμε γύρω από αυτά τα προϊόντα, γιατί θεωρούμε ότι αγοράζουμε ποιοτικά ε, εγχώρια προϊόντα, τα οποία πολλές φορές είναι μέτρια προϊόντα που δεν προέρχονται από εκεί που θα έπρεπε. Αυτό βεβαίως πλήττει και τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν προβάλλουν τόσο ποιοτικά προϊόντα και σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές και αυτό πλήττει την εικόνα των αυθεντικών προϊόντων. Για τα γεωργικά προϊόντα δεν υπάρχει θέμα γεωγραφικού σήματος, διότι από το 1992 προστατεύονται αυτά τα προϊόντα. Αλλά δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που ε, προστατεύει τα πολιτιστικά προϊόντα, τα αυθεντικά πολιτιστικά προϊόντα ή τα βιοτεχνικά προϊόντα. Γι' αυτό κάθε χώρα προσπαθεί να προστατεύσει αυτά τα μη γεωγραφικά προϊόντα με γεωγραφικό σήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει προστασία μη γεωγραφικών προϊόντων, το 2013 ε, χαρτογράφησε αυτές τις γεωγραφικές ενδείξεις για αυτά τα προϊόντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε ε, ενδεχομένως να έχουμε ένα ενιαίο γεωγραφικό σύστημα προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό απασχόλησε και την πράσινη βίβλο. 15 κράτη-μέλη έχουν προβάλλει ειδική προστασία, κάτι το οποίο όμως έχει πολλά κενά, διότι δεν καλύπτει όλη τη γεωγραφική Ευρωπαϊκή επικράτεια. Και υπάρχει και ετερογενής χαρακτήρας, διότι δεν υπάρχει σωστή προστασία με βάση τη γεωγραφική ένδειξη. Επίσης είναι άνηση αυτή η προστασία, διότι το κάθε κράτος μέλος ορίζει εγκάρσια μέτρα ή τομέακα και υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Αυτή η διαφορετικότητα είναι προβληματική για τις επιχειρήσεις που είναι πολύ μικρές, δηλαδή μιμιέψιλον. Ε. Θέλουν λοιπόν να εξασφαλίσουν τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες με υψηλό και ανυπέρβλητο κόστος. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις και για τις επιχειρήσεις και για τα εδάφη, συγκεκριμένα εδάφη και τους καταναλωτές για να υπάρχει ενιαία προστασία για την αξιοποίηση αυτών των προϊόντων προέλευσης για να καταπολεμήσουμε την παραχάραξη και να μην έχουμε τόσο υψηλό κόστος προστασίας. Έτσι οι μικροί βιοτέχνες θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να προσδιορίσουν αυτά τα προϊόντα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη μέσα στα πλαίσια μίας ε, συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, η γεωγραφική ένδειξη βοηθά για να βρεθούν τα μέσα και οι πόροι που δεν σχετίζονται μόνο με τους ε, άμεσους παραγωγούς. Πρόκειται για μια πολιτιστική δραστηριότητα και τουριστική, γιατί πρόκειται για τις περισσότερες φορές για αγροτικές ευάλωτες περιοχές. Επίσης, η γεωγραφική ένδειξη θα επιτρέψει μία ομοιογενή αναγνώριση αυτών των προϊόντων στην εσωτερική αγορά και θα δώσει και προστιθέμενη αξία σε αυτά τα προϊόντα. Έγινε μία έρευνα στον κλωστοϊφαντουργικό τομέα και είδαμε ότι όταν υπάρχει γεωγραφική ένδειξη υπάρχει προώθηση του προϊόντος κατά 25% περισσότερο. Επίσης, ο καταναλωτής ζητά μεγαλύτερη δυνατότητα ανείχνευσης του προϊόντος. Και αυτό που έχει σημασία είναι και η ποιότητα των προϊόντων ανάλογα με την προέλευσή τους. Είναι λοιπόν αναγνωρίσιμα προϊόντα και ο καταναλωτής θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική ένδειξη για να τα εμπιστευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραχάριξη, όμως μπορούμε να διαρθρώσουμε καλύτερα ένα μερίδιο της προσφοράς με βάση ομαδοποίησης προϊόντων από επαγγελματικούς κλάδους, με βάση και τους φυσικούς πόρους η εδαφική διαφορετικότητα δεν επιτρέπει τη ε, σωστή εντόπιση των γεωγραφικών ενδείξεων. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες ανησυχίες, να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα με καταγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χρειάζεται καταγραφή γιατί σχετίζεται με τα εμπλεκόμενα παράγωγα δικαιώματα και τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών. Στη συνέχεια αυτό το σύστημα σημαίνει ένα συγκεκριμένο κόστος το οποίο είναι περιορισμένο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίδοντας και στους καταναλωτές συγκεκριμένες εγγύσεις. Η πρωτοβουλία για γεωγραφική ένδειξη περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις για την δημιουργία γεωγραφικής ε, ένδειξης με βάση ε, βιβλία υποχρεώσεων ως προς τις παραγωγές και τις ε, καινοτομίες στον τομέα των, της βιοτεχνίας. Βεβαίως η γεωγραφική ένδειξη δημιουργεί ένα δεσμό μεταξύ του προϊόντος και της γεωγραφικής ένδειξης ανάλογα με την περίπτωση και τέλος το σύστημα θα πρέπει να προβλέπει την συνύπαρξη μεταξύ γεωγραφικών ενδείξεων και πνευματικών δικαιωμάτων. Η επέκταση αυτών των προϊόντων μέσα στα πλαίσια της προστασίας γεωγραφικής ένδειξης θα μας οδηγήσει στην προστασία της κληρονομιάς μας και θα βοηθήσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη για να δούμε κατά πόσο είναι μετρήσιμα όλα αυτά. Θα πρέπει να δούμε τι ισχύει με τις γεωγραφικές ενδείξεις στα αγροτικά προϊόντα. Στη Γαλλία, στον γαλακτοκομικό τομέα, έχουμε 2,8 το περισσότερη απασχόληση από τον ίδιο τομέα αν δεν τύχανε προστασίες με γεωγραφικές ενδείξεις. Αυτό ε, με βάση μία μελέτη και για το Ζαμπόν από την Μπαγιόν το 2008 έδειξε ότι χίλιες εργασίες επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν στις 3.000 που προϋπήρχαν, δηλαδή αύξηση της απασχόλησης κατά 30%. Γι' αυτό προτείνω το εξής χρονοδιάγραμμα. Η παρουσίαση της έκθεσης θα γίνει στις 20-21 Ιανουαρίου και στις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλλετε τροπολογίες. Θα τις εξετάσουμε στις 23 ή 24 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ φιλόδοξο θα έλεγα το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση. Θέλει κάποιος το λόγο. Δεν βλέπω ενδιαφέρον. Κύριος Καβαντά. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Θέλω όμως να πω ότι υποστηρίζω θερμά την προσέγγιση αυτή, γιατί σίγουρα δεν έχει την προστασία που θα έπρεπε ο τομέας αυτός, παρότι πραγματικά παράγει θέσεις εργασίας και παρέχει και σαφήνει για τον καταναλωτή κάτι που είναι για μας ιδιαίτερα πρόσφυλες. Στηρίζω λοιπόν τις προτάσεις της συγκήτριας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως ε, φαντάζομαι ότι ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σημείο αυτό. Το σημείο 26 της Μερίσιας Διάταξης έχει αναβληθεί, όμως έχουμε κάτι πολύματα από χθε και συγκεκριμένα τα σημεία 8 και 9. Ο κύριος Καβαντά έχει το λόγο ως εισηγητής. Θα είμαι πολύ ε, σύντομος κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για τα σύμφωνα συμβίωσης και τα περιουσιακά στοιχεία και την καταγραφή τους. Η κατάσταση έχει ως εξής. Μόνο συμβουλευτικό είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Το Συμβούλιο από μόνο του παίρνει τι αποφάσεις και προς το παρόν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας ως Κοινοβούλιο, τουλάχιστον στο πλαίσιο της πρώτης φάσης. Περιμένουμε λοιπόν την θέση του Συμβουλίου. Επειδή όμως ε, να μας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα γιατί είναι σημαντικό για πολλά άτομα και ιδίως ε, διαφορετικών εθνικοτήτων. Αποφασίσαμε να τονίσουμε ε, ότι το Συμβούλιο πρέπει να λάβει αποφάσεις ε, επί του θέματος αυτούς με ομοφωνία 25 χωρών όμως γιατί υπάρχουν τρεις χώρες που έχουν opt-out. Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο έχουν opt-out. Είναι λίγο εξωτική όλη η διαδικασία γιατί οι χώρε που έχουν opt-out συμμετέχουν παρόλα αυτά στη ζητήσει κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Πρόεδρο. Ε, ναι, έχετε δίκιο. Ε, ο κύριο Ντούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το θέμα αυτό σε ορισμένα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι βασικό να σεβαστούμε την επικουρικότητα. Δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-μέλη, καταχωρημένες ε, εταιρικές σχέσεις, σχέσεις ε, συντρόφων. Ε, Οπότε να έχουμε δεσμευτικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ένωσης για όλες τις χώρες, ακόμη και για τις χώρες όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ε, σχέσεις. Είναι λίγο περίεργο. Στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Ιταλία. Έχουμε ήδη θέματα τα οποία τα έχουν αναφέρει και η κυβέρνηση της δικής μου χώρας λοιπόν έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Οπότε θέλω να σημειώσετε ότι έχω επιφυλάξει για το θέμα αυτό. Γιατί θα ήταν πραγματικά αντιφατική κατάσταση κράτη ε, μέλη που δεν έχουν νομοθεσία για τέτοιες σχέσεις να ε, είναι υποχρεωμένες να την αναγνωρίσουν εάν έχει συναυθεί σε άλλη χώρα. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άλλη ερώτηση. Που παρακαλώ να απαντήσει ο κύριος Καβαντά. Η αρχή για τα θεμελιώδη δικαιώματα είπε ότι υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων. Για τις δυνατότητες δηλαδή που έχουν να επιλέξουν ε, είδος ε, σχέσεις τα ζευγάρια. Αντιμετωπίζει το θέμα το Συμβούλιο αυτό για να μην έχουμε διακρίσεις. Ούτως ώστε όλα τα ζευγάρια, ανεξάρτητα από το αν είναι παντρεμένοι ή έχουν καταχωρημένη σχέση συντρόφων, θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τον νόμο που προτιμούν. Από πλευράς Ιταλικής Προεδρίας ο κύριος Μπρούνο. Ο κύριος Καβαντά, κοιτάξτε να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Γιατί δεν ξέρω αν έχουν όλη την ίδια ενημέρωση. Η έκθεση εγκρίθηκε. Έχει ψηφιστεί. Το μόνο θέμα που θα μπορούσε... Ο, ο μόνος τρόπος να έχουμε περαιτέρω διευκρινήσεις είναι να ακούσουμε το Συμβούλιο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και καλημέρα σας. Η συζήτηση στο Συμβούλιο προωθήθηκε μέσα στα πλαίσια δύο ομάδων εργασίας. Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες όπως ε, ελέγχθηκε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα και ακαθόδη. Παρ' αυτά το Συμβούλιο, σε εργασίες μάλλον του Συμβουλίου υπήρχε αθρώα συμμετοχή θα προβούμε σε μία δήλωση του State of Play, της εξέλιξης κατάστασης, στις 4 ε, Δεκεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή. Ως προς τα ζητήματα που θίξατε, θα ήθελα να σας πω ότι τα προφίλ διακρίσεων που προαναφέρθηκαν σε σχέση με τους καταχωρημένους συντρόφους και τους συζύγους, οι διαφοροποιήσεις δεν υπάρχουν στα δύο νέα κείμενα, τα οποία επέβαλε η Ιταλική Προεδρία ως κείμενα συμβιβασμού, προσδίδοντας σημασία ότι και στις δύο προτάσεις υπάρχουν παράλληλες διατυπώσεις και άρθρα βεβαίως ε, τηρώντας τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στα δύο σχήματα, του συζύγους και τους ε, καταχωρημένους συντρόφους. Αυτό όσο αφορά το δικαιοδοτικό ζήτημα, καθώς και την επιλογή του νόμου που ισχύει στην κάθε περίπτωση. Άρα την ουσία δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των δύο κειμένων στο μέτρο του δυνατού. Έτσι έχουν εξελιχθεί οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι οι αποφάσεις ε, που αφορούν τα περιουσιακά δικαιώματα μεταξύ συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων είναι πολύ σημαντικά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Διότι με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερα ζευγάρια ζουν σε άλλες χώρες από τις χώρες στις οποίες έχουν συνάψει αυτές τις σχέσεις και υπάρχουν και ζευγάρια από διαφορετικές χώρες. Υπάρχουν 16 εκατομμύρια τουλάχιστον ζευγαριών και 650.000 εξ αυτών χωρίζουν κάθε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καθορίσουμε τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, να καθορίσουμε ποιο είναι το δίκαιο που πρέπει να εφαρμοστεί για τον διαχωρισμό των περιουσιακών τους ε, στοιχείων ζευγάρια ε, από διαφορετικό κράτος μέλος που χωρίζουν. Πρέπει να δουν λοιπόν ποιο είναι το δίκαιο, ποιο είναι το δικαστήριο που, στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν και υπάρχουν και μετά θέματα αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο να προσπαθεί να επιλέξει ο καθένας τη δικαιοδοσία που ε, τον βολεύει και δεν πρέπει επίσης να υπάρχει και αυτή η νομική αβεβαιότητα γιατί αυτό σημαίνει και υψηλότερο κόστος για να επιδιώξουν ε, τα ζευγάρια να καθορίσουν τα περιουσιακά τους δικαιώματα σε περιπτώσεις όχι μόνο χωρισμών αλλά και θανάτων. Πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να βασιστεί στα σχόλια και τις συστάσεις που έχουν ήδη γίνει. Συγκεκριμένα τα σχόλια που κάναμε για τον ε, κανονισμό Βρυξέλλες 1 για τις ε, κληρονομίες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται περιουσιακές επιπτώσεις αλλά όχι αναγκαία άλλες επιπτώσεις των καταχωρημένων, των καθεστώτων καταχωρημένων συντρόφων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να έχουν τέτοιο καθεστώς στην επικράτειά τους. Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο Συμβούλιο, διότι είστε λίγο ε, υπερβολικά διακριτικοί όταν συζητάτε κάποια ε, σημεία. Πρέπει να μας δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις. Δεν θα πρέπει ε, να έχετε μυστικά από την Επιτροπή μας. Και βλέπω ότι συμφωνεί και ο εισηγητή μα ο κύριος Καβαντά. Άρα, κύριε Μπρούνο, παρακαλώ, έχετε να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίε. Ευχαριστώ. Όπως ήδη είπα, θα προτιμούσα να το δούμε το θέμα λίγο αργότερα, όταν δούμε πού βρισκόμαστε σε δύο μέρες. Το Συμβούλιο θα συζητήσει τη θέση των μεμονωμένων κρατών μελών και των ζητημάτων που υπάρχουν στις ε, δύο αυτές περιπτώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να το αφήσουμε το θέμα μέχρι να συζητηθεί στο Συμβούλιο. Ο κύριος Μαρίνιου Επίντου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, δεν βρέθηκα χθε στη συνεδρίασή σας αλλά φαίνεται ότι παίζουμε το θέατρο των σκιών εδώ. Εδώ μιλάμε για ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Δηλαδή να μπορεί να επιλέξει τον ή την σύντροφο με τον οποίο θέλει να συζήσει. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει. Τώρα με αυτά τα καθεστώτα συζύγων ή καταχωρημένων συντρόφων, θα πρέπει να πω ότι εδώ υπάρχει το δικαίωμα της επιλογής. Εάν εγώ θέλω να συζήσω με έναν άνδρα, αυτό επίσης είναι θεμελιώδες δικαίωμά Θα πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά το θέμα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν ε, δεν μπορεί κανείς ε, να συζήσει επίσημα και καταχωρημένα ή να παντρευτεί όποιον θέλει. Και αυτό αφορά όχι μόνο τους ετεροφιλόφιλους, όπως ε, καταλάβατε. Θα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή και όχι από το τέλος. Ε, δηλαδή ο γάμος ε, δημιουργήθηκε για οικονομικούς, ε, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ως προς την εμβέλεια και το περιεχόμενό του. Το να μην επιτρέπουμε σε άτομα του ιδίου φύλου να μην μπορέσουν να καταχωρήσουν την συμβίωσή τους, αυτό παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Ο γάμος αφορά οποδήποτε, οποδήποτε, οποιοδήποτε θρήσκευμα. Στον, ε, Ισλαμισμό υπάρχει πολυγαμία, στην Καθολική Εκκλησία υπάρχει μονογαμία. Αλλά οποιοδήποτε μπορεί να διαλέξει το σύντροφο που επιθυμεί, ανεξάρτητα από το φίλο του. Δεν μπορούμε να παραβιάζουμε αυτό το θεμελιώδες δικαιώματα. Τώρα το συζυγικό καθεστώς διαφέρει. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι αυτή η θεμελιώδης, μάλλον αυτή η παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος. Ο άντρας μπορεί να παντρευτεί άντρα και γυναίκα γυναίκα δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο που θέλουν να μας επιβάλλουν. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα που δεν μπορούν να παραβιάζονται. Ε, Θέλετε το λόγο κύριε Καβαντά. Je vous remercie, euh, Président et Ευχαριστώ και καταρχάς σας ζητώ συγγνώμη γιατί νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσω ελαφρώς ε, σε αυτά που άκουσα. Καταρχάς να ζητήσω από την κυρία Ροζιέρε να κατοχυρώσει με δίπλωμα βρεσιτεχνίας ε, γεωγραφική ένδειξη ε, αυτό το χαρτομάνι, αυτό το τοίχο, το χάρτινο που κύριε Μπρούνο μόλις εσείς εφήβρατε, διότι άκουσα από την Ιταλική Προεδρία ουσιαστικά μια, κάτι που συνιστά πρόοδο. Είναι μια χώρα η οποία ασχολήθηκε με το σύνολο των ζητημάτων ε, που δείχνει ότι θέλει να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο σχεδόν 60 χρόνια μετά την εκκίνηση της ε, κοινής αγοράς που σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλη πρόοδο ότι αφορά τα οικονομικά, τα προϊόντα, τα πρότυπα, την υγεία κτλ. Όμως δεν καταφέρουμε οι τις ίδιες ελευθερίες να τις παραχωρήσουμε σε κάτι θεμελιώδες και πολύ σημαντικότερο από ε, ένα κιλό καρότα που περνάει τα σύνορα, όπως είπε ο συνάδελφος Μαρίνιο Πίντο και όπως είπε και πιο πριν η κυρία Χάουταλα. Δηλαδή, πρέπει να προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε τις ίδιες ελευθερίες για τον πληθυσμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε ίσως να σκεφτούν πιέσεις στα κράτη-μέλη που είναι επιφυλακτικά για να προχωρήσουν στην εναρμόνιση των δικαιωμάτων. Δεν είναι και κάτι το υπερβολικό. Δυσκολίες υπάρχουν, αλλά οι δυσκολίες υπάρχουν πάντα όταν θέλουμε να επιτελέσουμε πρόοδο και συμφωνώ μαζί σας. Όμως αυτή η προσέγγιση με απογοητεύει για το ρόλο ε, μια κυβέρνησης ε, την οποία περίμενα πολλά και που έχει ήδη παράσχει πολλά σε άλλους τομείς. Τελικά με τέτοιες συμπεριφορές δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι δημιουργούμε εμείς αυτούς τους ευρωσκεπτικιστές και αν είμαστε άκαμπτοι δεν θα ε, προχωρήσουμε. Πρέπει να έχουμε συγκρίσιμα ή εναρμονισμένα καθεστώτα. Αφήνουμε τον κόσμο να ε, περνά από τη μια χώρα στην άλλη. Δεν θα πρέπει να μπορεί να ζει και τον έρωτά του ένα ζευγάρι με ένα εναρμονισμένο καθεστώς. Πρέπει να δρομολογηθεί και αυτό. Δεν ξέρω αν θα το δρομολογήσει η Ιταλική Προεδρία το ζήτημα και οι χώρες που έχουν αυτή την ε, αυτοεξαίρεση θα έπρεπε να διαπραγματευτούν δεν μπορούμε τις μισές υποχρεώσεις ε, που πορεύουν από την, ε, ε, το γεγονό ότι ανήκουμε στον ίδιο χώρο να μην τις αφήσουμε να ισχύσουν. Θα πρέπει λοιπόν να μετακινηθούν οι αμετακίνητες μέχρι στιγμής κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρούνα, λέει ο πρόεδρος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω με δύο λόγια ως προς αυτά που είπε ο κύριος Καβαντά, μη με παρεξηγείτε. Οι εργασίες του Συμβουλίου οδήγησαν ε, σε πρόοδο σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν λίγους μήνες πριν. Υπάρχει ένα κείμενο συμβιβασμού που λαμβάνει υπόψη τη ευαισθητοποίησης των κρατών μελών. Πρόκειται για δύο ζητήματα που θα εγκριθούν με ομοφωνία. Το είπε και ο κύριος Καβαντά στην εισήγησή του. Όταν υπάρξει ομοφωνία θα γίνουν συνετά βήματα, όχι βεβαιασμένα, για να μην υπάρξουν υπαναχωρήσεις στις δύο προτάσεις. Υπάρχει λοιπόν μία σειρά διατάξεων που θα ε, διασαφινιστούν και από την Εθνική Ένωμη Τάξη. Μιλάμε για τις ε, διατάξεις αυτές και πώς μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο. Προσπαθούμε να μην υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των δύο αυτών διατάξεων και σχημάτων για να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες και τις λύσεις του γάμου ή της καταχώρησης αυτής συμβίωσης με βάση τους δύο κανονισμούς. Θα ήθελα λοιπόν να σας καθησυχάσω. Οι πιέσεις που επικαλεστήκατε κατά των πιο επιφυλακτικών κρατών έγιναν, γι' αυτό φτάνουμε στην τελική μορφή των δύο κειμένων που αποτελούν μια πολύ καλή βάση εργασίας έτσι ώστε να εγκριθούν και οι δύο κανονισμοί στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε εξαντλήσαμε τα θέματα της πρωινής μας συνεδρίασης και θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.